ε, ξαναρχίζει λοιπόν η συνεδρίαση, η οποία είχε διακοπεί στην προηγούμενη, στο τέλος της προηγούμενης ολομέλειας. Ε, τα πρακτικά ε, της ε, προηγούμενης συνόδου της 15ης Μαΐου του 2011 περιέχονται ήδη στο φάκελό σας. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, τα πρακτικά εγκρίνονται. Θα κάνω κάποιες, ένα, ε, ε, κάποιες παρατηρήσεις στο ξεκίνημα αυτής της ολομέλειας. Πρώτα απ' όλα, καλωσορίζουμε τον κύριο Αμούν Αλή Ραχμόν, πρόεδρο του Τατζικιστάν, ο οποίος ε, βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, σε επίσημη επίσκεψη. Przed chwilą spotkałem się z panem prezydentem, omawialiśmy Συνομίλησα με τον Πρόεδρο πριν από λίγο, αναφερθήκαμε στις διμερείς σχέσεις και βεβαίως μιλήσαμε και για τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητες στο Τατζικιστάν. Κυρίες και κύριοι, την 4η Ιουνίου ε, ε, είχαμε το γενέθλιο δύο σημαντικών γεγονότων. Το 1989 στις 4 Ιουνίου οι αρχές της λαϊκής Κίνας σταμάτησαν, έδωσαν ένα τέλος εις της των φοιτητών στην πλατεία Τιέναν Μέν. Όλοι θυμόμαστε το γεγονός αυτό. Την ίδια ημέρα πριν από τόσα χρόνια στην Πολωνία για πρώτη φορά ε, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έλαβαν χώρα ελεύθερες κοινοβουλευτικές εκλογές και τα μέλη της ε, αντιπολίτευσης, της δημοκρατικής αντιπολίτευσης ε, κέρδισαν και πήραν σχεδόν όλους τους, όλες τις έδρες. Οι εκπρόσωποι της δημοκρατικής αντιπολίτευσης